του Προέδρου. Το Συμβούλιο ζήτησε την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 154, της διαδικασίας του κατεπήγοντος, για την εξής πρόταση. Πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου για αλλαγή του κανονισμού υπαριθμών 1150 του 2000 για εφαρμογή της απόφασης 2007 436 Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των κοινοτήτων. Ένας πάρα πολύ ωραίος τίτλος, πίσω από τον οποίο υποκρύπτεται ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα. Δηλαδή, με ποιον τρόπο συνεισφέρουν οι χώρες στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Η ψηφοφορία ε, επί του αιτήματο αύριο το πρωί στις 9. Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του κανονισμού, ο πρόεδρος της διάσκεψης των Προέδρων με ενημέρωση για το εξής. Δεν υπήρξαν κάποιες